ενεργειακής αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας μάλλον, δίνω το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά, τον κύριο Ταμπουράνο. Doesn't work. Yes, okay. Okay. Καλησπέρα, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το ενεργειακό σήμα είναι μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχία που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια και το έχουν αντιγράψει πάρα πολλέ χώρε στον κόσμο. Είναι ένα είδο ενεργειακού διαβατηρίου που γνωρίζουν οι πάντε και εγγυάται ότι όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στο σπίτι των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων έχουν συγκεκριμένε πληροφορίε όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και όσον αφορά άλλα θεμελιώδη χαρακτηριστικά. Μαζί με τον οικολογικό σχεδιασμό, το ενεργειακό αυτό σήμα επέτρεψε μέσα σε λίγα χρόνια στου Ευρωπαίου πολίτε να μπορούν να αγοράσουν πλυντήρια, ψυγεία, φούρνου, λαμπτήρε, ε, λέβητε οι οποίοι είναι όλο και πιο ενεργειακά αποδοτικοί, έχουν μειωμένε βλαβερέ συνέπειε, καθώ επίση και μειωμένε εκπομπέ. Κατά αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι ασθένειε, μειώνονται οι βλαβερέ συνέπειε στο περιβάλλον και επίση μειώνεται και η πολιτική εξάρτηση και η ενεργειακή εξάρτηση τη υπήρου μα. Εδώ και κάποια χρόνια όμω οι πληροφορίε ετικέτα αυτή δεν είναι τόσο αποδοτικέ, θα λέγαμε. Οι καταναλωτέ συγχύσονται αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να καταλάβουν πάρα πολύ καλά πώ λειτουργούν οι τόσο διαφορετικέ κλίμακε και διαφορετικέ κατηγορίε, διαφορετικέ βαθμίδε και τι σημαίνει τελικά αυτό και κάθε προϊόν όσον αφορά την κατανάλωση ενέργεια και την τιμή του. Ήρθε λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε τον ενεργειακό αυτό διαβατήριο πιο αποτελεσματικό, να τον ανανεώσουμε και να αποφεληθούμε από τα ωφέλη τη ψηφιακή τεχνολογία. Πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να καταφέρουμε να απευθυνθούμε στην υφιστάμενη και μελλοντική αγορά. Κατά τη σύνταξη της ε, έκθεσης αυτής ε, προσπάθησα να θέσω κάποιους στόχους. Είπα ότι θα πρέπει να βάλουμε μια τάξη λίγο στα πράγματα, να καταργήσουμε όλα αυτά τα σύντα που βλέπουμε δίπλα σε διάφορες κατηγορίες, να καταστήσουμε το σήμα πιο ψηφιακό και να έχουμε επίσης και καλύτερη εποπτεία της αγοράς. Άκουσα τι είχαν να πει ο κλάδος, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εποπτικές αρχές, οι ίδιοι έμποροι, οι αρχές τυποποίησης, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά και οι ίδιοι πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν σε διάφορα πολιτικά κινήματα. Πρότεινα λοιπόν μια έκθεση ιδιαίτερα ευρεία και συνθετική προκειμένου να καταφέρουμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών μετά το σκάνδαλο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και να αυξηθεί κατά αυτόν τον τρόπο η εξοπιστή οποιασδήποτε νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ελπίζω ότι πραγματικά θα οδηγηθούμε σε μια νέα μοντέρνα ψηφιακή ετικέτα, θα την αποκαλούσε ετικέτα 2.0 και Ελπίζω ότι η ετικέτα αυτή θα αποτελέσει επίση και την αρχή για τη δημιουργία μια βάση δεδομένων για όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά, τα οποία ο κάθε πολίτη θα μπορεί να συμβουλεύεται στη δική του τη γλώσσα. Προσπάθησα λοιπόν στα πλαίσια της έκθεσης αυτής, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Βιομηχανίας, να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα το οποίο ελπίζω ότι και όλοι οι ολομέλοι εδώ πέρα την Τετάρτη θα δεχθεί με τον ίδιο ενθουσιασμό. Μέσα στι βελτιώσει που βλέπουμε στο κείμενο αυτό, θέλω να τονίσω τι ακόλουθε. Πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχύσει το μηχανισμό του ορισμού των προτύπων και της ξεχωριστή ταξινόμηση που έχουμε με βάση τι ενεργειακέ κατηγορίε. Χρειάζεται καλύτερο λοιπόν έλεγχο, ο οποίο θα συνάδει με, το, με την πραγματική χρήση των προϊόντων. Όλε οι δοκιμέ θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά και θα πρέπει τις πληροφορίες αυτές να τις έχουν όλες οι αρχές εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε επίση ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που να έχει δύο τμήματα. Ένα δημόσιο τμήμα και ένα τμήμα το οποίο θα είναι μόνο για τις αρμόδιες αρχές. Μια τέτοια βάση δεδομένων για τα προϊόντα θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό και θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο ψηφιακό κώδικα πάνω στην ετικέτα που θα επιτρέπει στον οποιονδήποτε να γνωρίζει ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος. Είπαμε επίση ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα αυτόματο μηχανισμό προκειμένου να καταργηθούν όλα αυτά τα θετικά πρόσημα τα οποία έχουμε σε διάφορε κατηγορίε, όπω για παράδειγμα α-συν, α2-συν, α3-συν, πρέπει αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό με εξαίρεση μόνο του λέβητε που παρουσιάζουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και του οποίου χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για να γίνει αυτή η κατάργηση. Είπαμε επίση ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα γενικότερο κανόνα όσον αφορά την αναπροσαρμογή τη κλίμακα, ιδίω όσον αφορά τι ανώτερε κατηγορίε Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό, Σε ζητώ συγγνώμη. Είχατε τέσσερα λεπτά. Πρέπει να παραμείνετε πιστό στο χρόνο που σας έχετε δοθεί. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, δεν θέλω να σας διακόψω, <clears throat> αλλά σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο <clears throat> αγόρευσης. Και επίσης είναι συνηθισμένο όταν μιλάτε να είστε όρθιος, να είστε είναι τμήμα της κοινοβουλευτικής παράδοσης. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μέλμστρουμ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. <coughs> Θέλω καταρχήν να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον κύριο Ταμπουράνο, τον εισηγητή και τους ισχυροδησηγητές για το πάρα πολύ σημαντικό τους έργο μία από τις βασικές υποβόσκουσες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει τη δυνατότητα επιλογής στους καταναλωτές και να οδηγήσουν αυτή την πορεία προς την καθαρή ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στα πλαίσια αυτά, τον Ιούλιο του 2015 η Κομισιόν έκανε μια πρόταση αναθεώρησης και επικαιροποίησης του πλαισίου για τη σήμανση ενεργητικής αποδοτικότητας. Αυτή η σήμανση έχει εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν πιο ευφυείς επιλογές που θα εξοικονομήσουν χρήματα και ενέργεια. Πάνω από 50% ελέγχουν την ενεργειακή απόδοση που αγοράσουν ένα καινούργιο πλυντήριο ή ένα καινούργιο ψυγείο. Οι πολιτικές αυτές οδηγούν σε σημαντικές εξοικονομήσεις που φτάνουν περίπου τα 465 εκατομμύρια ευρώ και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 55 δισεκατομμύρια πρόσθετο τζίρο για τις επιχειρήσεις ε, που παράγουν τέτοια ε, προϊόντα. Οπότε αυτό είναι και θέμα και ανταγωνιστικότητα και όχι μόνο εξοικονόμησης ενέργειας. Όλη αυτή η διαδικασία έχει οδηγήσει σε όλο και πιο αποδοτικά ενεργειακά προϊόντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε. Αλλά βέβαια και αυτή η σήμανση είναι θύμα τη επιτυχία τη. Πρέπει να αλλάξουμε τη σήμανση, γιατί τα περισσότερα προϊόντα βρίσκονται στις πιο ψηλέ κατηγορίες και έτσι δεν υπάρχει απαραίτητη διαφοροποίηση για τους καταναλωτές. Όπως είπε ο εισηγητής, <clears throat> είναι σχεδόν όλα τα προϊόντα στην κατηγορία α, α α2 σ α3 σ α νη σίγμα. Και με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές θα κάνουν σωστή επιλογή. Μετά από πολλές λοιπόν διαβουλεύσεις και μετά από αιτήσει των καταναλωτών, η Κομισιόν προτιμά να επανέλθουμε στην αρχική κλίμακα από το A ω το G λατινικό για την ενεργειακή απόδοση, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δώσουμε σαφείς πληροφορίε στους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να κάνουν τις σωστές και καλά πληροφορημένε αποφάσεις. Σήμερα οι καταναλωτές πρέπει να ξέρουν για την ενεργειακή απόδοση των συσκευών, όπω θέλουν να ξέρουν για τις χίλιο θερμίδες στα τρόφιμα τα οποία τρώνε. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε την θέληση του εισηγητή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας έχει βοηθήσει να κάνουμε σημαντική πρόοδο σε αυτή την πρόταση. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες <clears throat> που περιέχονται στην έκθεση όπως η αναπροσαρμογή των κλιμάκων αλλά υπάρχουν δύο προτάσεις που αναφέρονται στην πρόταση αυτή που εμείς φοβόμαστε ότι μπορούν να υποσκάψουν και την επιτυχία του σχεδίου μας για την ενεργειακή σήμανση. Πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων αυτή τον αντίκτυπό τους. Το να κρατούν οι, οι, οι κατασκευαστές αυτών των, των ε, συσκευών στοιχεία για όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία, που θα είναι πληροφορίες προσβάσιμα από μια κεντρική βάση, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε ρεαλιστικό, όπως και το να υπάρχει μια τράπεζα δεδομένων μέσα σε ένα χρόνο και όχι σε δύο. Η βιασύνη θα οδηγήσει σε κακή ποιότητα δεδομένων <clears throat> και σε άχθος για του κατασκευαστέ. Μπορεί να, μην, μπορεί να επιτευχθεί καν αυτή η προθεσμία. Εγώ προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναπροσαρμογή τη κλίμακο ώστε να εφαρμοστούν όλα αυτά το ταχύτερο δυνατόν χωρί μεγάλο διοικητικό άχθο. Θα πρέπει η νέα σήμανση να εξυπηρετεί του καταναλωτέ. είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν οποιαδήποτε αλλαγή και πρέπει να του βοηθήσουμε να συνεχίσουν να το πράττουν αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο. Και τώρα έρχονται οι ομιλητές εκ των πολιτικών ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Ρόιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την ε, καλή συνεργασία και κουραστική θα έλεγα. Δεύτερον, η ετικέτα είναι μια επιτυχία, το είπαν όλοι οι συνάδελφοι. Πετύχαμε ένα συμβιβασμό με, με πολλή δουλειά. Και θέλω να πω πως αν αλλάξει ο συμβασμός αυτό στην ψηφοφορία την Τετάρτη, ε, δεν θα τον δεχτούμε. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν το εάν αξίζει να υποβάλουμε τροπολογίες ή να αφήσουμε τα όσα πετύχαμε στην Επιτροπή με τα υπέρ και τα κατά να μείνει ως έχει. Να πω δύο μεγάλες επιφυλάξεις. Η πρώτη αφορά την ε, τράπεζα δεδομένων. Ε, υποτίθεται ότι ασχολούμαστε με τα σοβαρά και τα μεγάλα και οι κυβερνήσεις πραγματικά δεν συνεργάζονται για σοβαρά κεντρικά ευρωπαϊκά ζητήματα. και η έκθεση αυτή η οποία η έκθεση δοκιμής η οποία θα πάει υποτίθεται στην ε, βάση δεδομένων τι σημαίνει, δηλαδή θα πρέπει για 25.000 προϊόντα που έχει ένας μέσος κατασκευαστής να υποβάλει 25.000 εκθέσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το κόστος, η Κομισιόν μιλάει για αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, γύρω στα 28, εμείς υποθέτουμε ότι θα είναι ακόμη περισσότερα. Και οπωσδήποτε οι εποπτικές αρχές ε, δεν ενδιαφέρονται και δεν θέλουν πραγματικά όλον αυτό τον όγκο της δουλειάς. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε κάποια λογικά δεδομένα και να μην ξεχνάμε ότι είναι και πολύ ευαίσθητα. Εγώ με το δικό μου το χρονόμετρο έχω δύο λεπτά ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Ενάμιση λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Δύο λεπτά, λέει ο κύριος Ρόιλ. Όχι, συγγνώμη, ενάμιση γράφει εδώ. Συγγνώμη, σε έδωσα και παραπάνω από 1,5 λεπτό σας έδωσα και 20 δευτερόλεπτα τζάμπα. Από τη σοσιαλιστική ομάδα λοιπόν. Η κυρία Μαρτίνα Βέανα. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή καθώς και όλους τους συναδέλφους που όπως ο κύριος ε, Ρόιλ ε, ήδη έχει ευχαριστήσει για την πολύ καλή συνεργασία. Ένα βασικό στοιχείο, ένα ακρογωνιαίο λήθο τη Ενεργειακή Ένωση είναι η ενεργειακή απόδοση. Με την καλύτερη χρήση τη ενέργεια μπορούμε να κάνουμε σημαντικέ εξοικονομήσει και έτσι έχουμε ένα πολύ μεγάλο δυναμικό για να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση και έτσι να βοηθήσουμε και την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή. Αυτό όμω σημαίνει ότι και η η ενεργειακή απόδοση οδηγεί και σε μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τρίτες χώρες και μεγαλύτερη δυνατότητα για τις επιχειρήσεις. Με την αναδιάταξη των τάξεων, των κατηγοριών ε, ενεργειακής απόδοσης θα μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη, θα μπορούν οι να κάνουν μια καλύτερη σύγκριση και να αγοράζουν εν γνώση τα καλύτερα προϊόντα. αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τροποποιηθεί η, η κατάταξη ώστε να μπορέσει να συνεχίσει η πρόοδος η οποία γίνεται για την ενεργειακή απόδοση. Όλα αυτά είναι προς το συμφέρον της βιομηχανίας γιατί αυτό θα οδηγήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Σήμερα λόγω της επιτυχίας της βιομηχανίας είναι πάρα πολλά τα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στις ανώτερες ταξι, ε, αποδοτικότητα και είναι πολύ λίγα τα οποία βρισκόνται στις χαμηλότερε κατηγορίε. Αυτό οδηγεί σε αυξανόμενη σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών. Είναι καιρό να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη σαφήνεια σε ό,τι αφορά την αγορά ηλεκτρικών συσκευών και να κατανοούν καλύτερα οι καταναλωτέ τι σημαίνουν οι σημάσει αυτέ. Γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορέσαμε όλοι μαζί να καταλήξουμε σε μια εποφελή συμβαστική λύση για τα περισσότερα προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι επανερχόμαστε σε μια ενιαία κατάταξη από το α ως το g λατινικό για όλα τα προϊόντα. Επομένω ο καταναλωτής με μία ματιά θα μπορεί να συγκρίνει όλα τα προϊόντα και να ξέρει ποια είναι πιο αποδοτικά. Δεύτερον, είναι καλό ότι τα πιο, πιο συνηθισμένα ε, πιο συνδυσμένες ηλεκτρικές συσκευές μέσα σε 21 ε, μήνες θα μπορέσουν να εφοδιαστούν με το νέο σύστημα, εκτός από ορισμένε συσκευέ θέμας που θα χρειαστούν πέντε χρόνια. Έτσι θα υπάρχει και η δυνατότητα για τις ε, ε, δημόσιες αρχές να υπάρχει μια εποπτεία της αγοράς με μια βάση δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία αυτών των προϊόντων. Και αυτό μπορεί να είναι θετικό και για τα κράτη-μέλη. Από εμάς ως σοσιαδημοκράτες υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα. Εμεί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια κεντρική τράπεζα δεδομένων και όσοι Σοσιαλδημοκράτε θεωρούμε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δώσουν κίνητρα στου καταναλωτέ χαμηλών εισοδημάτων. Με όλε αυτέ λοιπόν τι συμβαστικές λύσει, νομίζω ότι έχουμε πετύχει το στόχο μα και αυτή η απόφαση μπορεί να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστούμε και τον εισηγητή για τι προσπάθειές του. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Κυρία Βέρνερ, από την ομάδα ECR, ο βουλευτή κύριο Άσλι Φόξ. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δική μου πολιτική ομάδα είναι υπέρ τη έκθεση αυτή για την ενεργειακή απόδοση και τη σήμανση. Όντω, προκαλείται σύγχυση αυτή τη στιγμή στου καταναλωτέ με το φυστάμενο σύστημα και χαίρομαι πάρα πολύ ότι οι κατηγορίε ΑΣΥΝ, α 2 α προκειται να καταργηθούν και θα χρησιμοποιήσουμε την κλασική κλίμακα Α έω G. Χαίρομαι πάρα πολύ που προβλέπεται επίση μια πενταετή περίοδο προκειμένου να γίνει αυτή η μετάβαση. Είναι λογική αυτή η χρονική περίοδο και για του καταναλωτέ αλλά και για του παραγωγού. Παρ' αυτά, έχουμε κάποιε επιφυλάξει όσον αφορά τη δημιουργία κεντρική τις δεδομένων. Είμαστε όμως ικανοποιημένοι που το προτινόμενο κείμενο πραγματικά δείχνει ποιε ήταν απαιτήσει για τους παραγωγούς, κάτι που δεν υπήρχε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η βάση αυτή δεδομένων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο υποπτήρες αγοράς, δεν θα θέλαμε όμως να αποτελέσει βάρος και άρθος για τον ε, κλάδο. Επίση, χαιρόμαστε που η έκθεση αυτή ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλογιστεί αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια μεταβατική περίοδο 10 ετών προκειμένου να προχωρήσουμε στην αναπροσαρμογή τη κλίμακα στι ενεργειακέ κατηγορίε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο αυτό προκειμένου να αυξήσουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εν γέννη, θεωρούμε ότι η νομοθεσία αυτή θα υποφελήσει του καταναλωτέ χωρί να δημιουργεί περαιτέρω δαπάνε Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει σωστά στην πράξη και είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε κάποιε τροπολογίε άλλων πολιτικών ομάδων που κάνουν το σύστημα πάρα πολύ αυστηρό και δεν θα λειτουργήσουν υπέρ του όλου συστήματο και σίγουρα όχι υπέρ των επιχειρήσεων. Εν γέννη πάντω είμαστε υπέρ τη πρόταση αυτή και θα την υπερψηφίσουμε την Τετάρτη. Ευχαριστώ. Κύριε Φόξ, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Σάνι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε, έχετε αναφερθεί στο νέο σύστημα για τα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος, αυτά τα οποία βοηθούν καλύτερα τον καταναλωτή, ότι μπορεί να διακρίνει καλύτερα τις διαφορές μεταξύ των ε, προϊόντων ο καταναλωτής, αλλά Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για την ε, βιομηχανία. Μήπως πρέπει να υπάρχει μια προστασία και για τη βιομηχανία. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, όντως τα σήματα αυτά θα βοηθήσουν τους καταναλωτές. Έχουμε κάποιες κατηγορίες ε, προϊόντων όπου έχουμε α συν, α2 συν, α3 συν τα λιγότερα αποδοτικά έχουν το ΑΣ. Ο καταναλωτή νομίζει ότι αγοράζει ένα ενεργειακά αποδοτικό προϊόν, το οποίο όμω στην πραγματικότητα δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό. Και προφανώ μπορεί το σύστημα αυτό, το εφιστάμενο σύστημα, να αποτελέσει άχθο για τη βιομηχανία και να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστο για του καταναλωτέ. Η συγκεκριμένη όμω πρόταση πετυχαίνει την κατάλληλη ισορροπία. Thank Βίρινγκ από την ομάδα του Δύο λεπτά. Ehm, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η μεταρρύθμιση της ετικέτας πρέπει να επιτύχει δύο στόχους. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να παρακινήσουμε τους παραγωγούς σε περισσότερη καινοτομία για να φέρει καλύτερες συσκευές στην αγορά. Δεύτερον, θέλουμε να έχουμε καλύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω καλύτερης συνεργασίας ε, των εποπτικών υπηρεσιών. Τέλος, θα πρέπει να φροντίσουμε ο καταναλωτής να μπορεί να αγοράζει πιο οικονομικές συσκευές. Έτσι μειώνεται η κατανάλωση και πέφτει ο λογαριασμός του ηλεκτρικού. Είναι σημαντικό λοιπόν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο με έναν τρόπο ο οποίος θα βοηθάει και τον καταναλωτή και τους παραγωγούς ε, και τους χρήστες. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουν υπόψη και τους μικρούς ε, αντιπροσώπους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν πρέπει να επιβαρυνθούν ιδιαίτερα. Και από αυτοί συνάδελφοι θεωρώ ότι με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή έχουμε μια ισορροπία και ένα καλό συμβιβασμό μεταξύ των θέσεων των πολιτικών ομάδων και των ενδιαφερομένων. Θεωρώ ότι επιλέξαμε μια φιλόδοξη προσέγγιση που ξεκαθαρίζει σε όλους το τι επιτρέπεται και το τι όχι. Και το τι γίνεται και το τι όχι. Είμαστε ακόμα στα απόνερα του σκανδάλου της Volkswagen. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του ο καταναλωτής στις διάφορες ετικέτες που βλέπει. Και θέλω να είμαι ξεκαθαρή, ένα ψυγείο το οποίο καίει περισσότερο ρεύμα είναι για μένα εξίσου άσχημο με ένα αυτοκίνητο που καίει περισσότερο δίζελ. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε παραπλάνηση του καταναλωτή, βλάβη του περιβάλλοντος και θα το νιώσουμε και στο πορτοφόλι, είτε στην αντλία είτε στο λογαριασμό του ρεύματος. και θα υπερασπιστώ αυτή την φιλόδοξη προσέγγιση που έχουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Βίρινγκ για την Γκουε. Ο κύριος Σιλικιώτης έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον Τάριο Ταμπουράνο για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Η ομάδα μας η ΚΟΥΕ υποστήριξε εξ αρχής πως είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ένα σύστημα ενεργειακής επισήμασης ευνόητο στους καταναλωτές το οποίο όμω να περιλαμβάνει και όλε τι απαραίτητε πληροφορίε. Χαιρετίζομαι λοιπόν τι προτάσει που περιλαμβάνονται στην έκθεση για διαγραφή των παραπλανητικών συμβόλων και μετάβαση σε ένα απλούστερο ενιαίο σύστημα ανεπισήμανση από το A ε ως το g. έτσι οι καταναλωτέ θα έχουν σαφέστερε ενδείξει για την ενεργειακή απόδοση ενό προϊόντο και θα, είναι σε θέση να κάνουν συνειδητέ επιλογέ με τι οποίε θα εξοικονομούν ενέργεια αλλά και χρήματα γι' αυτό και καταθέσαμε σχετική τροπολογία ζητώντας να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό άμεσα και σε όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα. εξίσου σημαντική είναι και η πρόταση που προωθείται στην έκθεση για δημιουργία μιας νέας ψηφιακής βάσης δεδομένων για τα προϊόντα στην οποία οι καταναλωτές θα έχουν δωρεάν πρόσβαση. ωστόσο θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό η βάση αυτή να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα αλλά και για τα δικαιώματα των καταναλωτών ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να τεθεί έτσι φραγμός στην εσχροκέδρια και στην παραπλάνηση των καταναλωτών από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για να μπορέσουμε όμως να προχωρήσουμε σε όλα αυτά είναι σημαντικό να δώσουμε όλοι ψήφο εμπιστοσύνη στον εισηγητή ώστε να αρχίσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Uh, Εξ ονόματος των Πρασίνων, ο κύριος Γιαβόρ έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση που διεξάγουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήταν της μεγαλύτερης σημασίας λοιπόν να είναι καλά πληροφορημένοι όλοι οι καταναλωτές σε σχέση για την ενεργειακή απόδοση και κατανάλωση των συσκευών που χρησιμοποιούν. Αλλά η, επιτρο... η έκθεση που εγκρίναμε στην Επιτροπή Ήτρε δεν είχε πολλά στοιχεία από το αρχικό περιεχόμενο του κυρίου Ταμπουρίνο. Δεν είναι θετικό να έχει ο εισηγητής μία ε, εντολή για τον τρίλογο που λέει ότι όλα τα προϊόντα από το 2020 θα πρέπει να έχουν μια ετικετοθεσία, μια σήμανση από το α ως το g. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι όμως ο, ο κατανοητής να έχει μια πληροφόρηση για την χρησιμοποίηση της ενέργειας κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Και αυτό χρειάζεται μια ενιαία αντιμετώπιση. Ευχαριστώ για την ομάδα ENF η κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, η έκθεση αυτή για σήμανση ενεργειακή των συσκευών είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον ε, καταναλωτή και όπως είπε και ο συγητής υπάρχει μια νέα σαφέστερη ε, σήμανση. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της ε, Τράπεζας Δεδομένων που είναι ένα αμφιλεγόμενο, περισσότερο αμφιλεγόμενο θέμα για το αν θα κάνει πιο σαφή και πιο εύκολη την εργασία των ε, κρατικών αρχών. Η καλύτερη σήμανση, η χρήση μιας κλίμακος από το α στο g, κάνει πιο απλή την αντιμετώπιση την, ε, ε, των προϊόντων αυτών από τον καταναλωτή, γιατί ο καταναλωτής τώρα τα έχει χάσει με, με τη σήμανση που φτάνει στο α με 3 συν. 85% των καταναλωτών τώρα δίνουν σημασία σε αυτό το οποίο αναφέρει η ετικέτα στα προϊόντα τα οποία αγοράζουν και αυτό είναι κάτι το οποίο προωθεί και την ε, καινοτομία στην ε, παραγωγή αυτών των προϊόντων και φυσικά και στην ενεργειακή εξοικονόμηση. Είναι απαραίτητο όμως να υπάρξει αυτή η ενία αντιμετώπιση από το α ως το g και έτσι με το να αγοράσουν τα πιο αποδοτικά προϊόντα οι καταναλωτές μειώνεται και η χρήση ενέργειας και μειώνεται και το κόστος των προϊόντων αυτών. Θα πρέπει να γίνεται όμως η μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης κατά πραγματικές συνθήκες και όχι σε ειδικέ συνθήκες. Αν λοιπόν υπάρξει ένα προϊόν το οποίο βρίσκεται στην πολύ ψηλή κατηγορία, να, όταν πάρα προϊόντα στις ψηλές κατηγορίες θα πρέπει να προσαρμόζεται αυτόματα η κατηγοριοποίηση. Αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Ο κύριος Γκούναρ Χουκμαρκ. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ να ευχαριστήσω και τον εισηγητή τον κύριο Ταμπουράνο. Κάθε φορά που μιλάμε για επισήμανση ενεργειακή απόδοση, δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο κατά νου ότι πρέπει να θέσουμε τα πράγματα σε μια σωστή βάση αλλά σε μια βάση που θα είναι όλο και καλύτερη, όλο και πιο βελτιωμένη. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο, σαφέ σύστημα επισήμανση που θα γίνεται ευκόλω κατανοητό από τους Ευρωπαίους πολίτες. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα κάνουν τις καλύτερες επιλογές και θα επιλέγουν τελικά τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούν καλύτερες τεχνολογίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη συζήτηση που κάνουμε εδώ, αλλά και για τη συζήτηση που κάνουμε εν γέννη για τη χρήση της ενέργειας και σε, άλλες, σε άλλους χώρους. Για οποιαδήποτε συσκευή και αν μιλάμε, κάθε νέα μορφή της πιο εξελιγμένη μορφή της είναι καλύτερη από παλαιότερη μορφή της. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παγώσουμε τη διαδικασία αυτή της τεχνολογικής εξέλιξης των προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην εστιαζόμαστε πάρα πολύ στην γραφειοκρατία. Δεν νομίζω ότι μπορούμε μέσω γραφειοκρατίας ή μέσω νέων κανονισμών να πετύχουμε αυτή την ευκταία πρόοδο. Αν λοιπόν αυτή η περίφημη βάση δεδομένων δεν είναι απλή και μη γρεφοκρατική, τότε πραγματικά θα παγώσει οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη, δεν θα βοηθήσει να πετύχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει μια έντονη σχέση με του επιχειρηματίε εδώ πέρα και ότι θα πρέπει στη βάση των αποφάσεών μα να έχουμε και τη συμβολή των επιχειρηματιών. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Φλάβιο Τζανονάτο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κλιματική αλληλή αλλά και το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης και ασφάλειας έχουν να κάνουν με τις σωστές επιλογές των καταναλωτών, οι οποίοι επιλέγοντας συσκευές τελικά πιο αποδοτικές από ενεργειακής πλευράς ουσιαστικά οδηγούν σε μια εξοικονόμηση της ενέργειας όπου θα φτάσει τα 170 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου σε εξοικονόμηση μέχρι το 2020. Καταλαβαίνετε ότι η κατανάλωση αυτή τη στιγμή, ιδίω σε χώρε όπω η Ιταλία, είναι τεράστια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή οικιακών συσκευών που θα είναι ενεργειακά αποδοτικέ. Και θα πρέπει όμω παράλληλα οι Ευρωπαίοι πολίτε να πλησιώνονται από τι κατάλληλε κοινοτικέ πολιτικέ για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντο. Το κείμενο λοιπόν αυτό είναι θετικό. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ταμπουράνο για την εξαιρετική του έκθεση και συμφωνούμε με την έκθεση αυτή. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει ο κύριος Ταμπουράνο λέγοντας ότι υπάρχει μια έντονη τεχνολογική εξέλιξη, ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς την νέα αυτή ε, τεχνολογική εξέλιξη, δημιουργώντας ένα σύστημα βαθμίδων και κατηγοριών που θα γίνεται πολύ πιο εύκολα κατανοητό από τους Ευρωπαίους πολίτες. Ελπίζω λοιπόν ότι με βοήθεια του Συμβουλίου θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποια κοινά σημεία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πλάνκο Λόπες έχει το λόγο. Ήδη όπως αναφέρθηκε έχουμε αυτόν τον κανονισμό για την ετικετοθεσία όσον αφορά την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα. Και θα πρέπει να ενημερώνεται ο πεολίτη ή ο καταναλωτή τέλο πάντων για να μπορεί να ξέρει ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιε είναι οι επιπτώσει κάποιων προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά και μπορούν να έχουν όσον αφορά το ηλεκτρικό, το ενεργειακό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα δεν πρόκειται για έναν κανονισμό ο οποίος πρόκειται να μας βοηθήσει να πετύχουμε τον στόχο της μείωσης των εκπομπών. Οπότε και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δούμε τι θα γίνει με αυτή την επισήμανση ε, για να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη αποδοτικότητα διαφόρων προϊόντων και θα πρέπει να υπάρξει η κατηγοριοποίησή τους ε, ανάλογα με το τι, τι προσφέρουν. Ε, να δούμε τι γίνεται και με την βιομηχανία της θέρμανσης γιατί και εκεί πέρα τώρα μπήκαν τέτοιες επισημάνσεις και από την άλλη μεριά επίσης αυτή η κατηγοριοποίηση θα μας γλιτώσει από κάποιες περιπτώσεις όπως DDA ε, για να χρησιμοποιούμε κάποιες, ε, κάποια προϊόντα του εργαστηρίου. Τι ήταν αυτό. Ε, Και τώρα ο κύριος Κόφουντ έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε. Οι αποφάσεις ελήφθησαν από το 2010 και τώρα. Θέλουμε μέχρι το 2020 να έχουμε εξοικονόμηση ενεργείας όσο είναι η ενέργεια που καταναλώνει όλη η Ιταλία και επίσης έχουμε ε, εξοικονόμηση περί τις 3.000 ε, κορώνες ετησίως. Όλα αυτά για τους Ευρωπαίους πολίτες είτε προέρχονται από την Τσεχία, είτε προέρχονται από τη Δανία, την Πορτογαλία, οπότε έτσι πιστεύω ότι θα ε, πετύχουν μια σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία και ε, δεν έχουμε το α, συν, α, συν, συν, συν και όλα αυτά τα οποία τόσο έφεραν τη σύγχυση σχετικά με τα πλυντήρια, της ηλεκτρικές σκούπες κλπ. Γιατί στο μέλλον θα έχουμε την βαθμονόμηση από το α μέχρι το g, πιο εύκολο αυτό, θα ωφεληθεί το περιβάλλον και θα ωφεληθεί και η τσέπη μας στον πρώτο λογαριασμό της ΔΕΗ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Και τώρα, κάτσε διάει ο πρώτος, ο κύριος Μπόγκοβιτς, έχετε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ στηρίζω αυτή την ε, πρωτοβουλία για να επιτύχουμε πρόοδο και αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας βεβαίως αποκρίνεται και στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης και τα λοιπά τα τελευταία 20 χρόνια η Ευρώπη ασχολείται εντατικά με αυτό το θέμα και από ό,τι φαίνεται έχουν τελειώσει τα συν για να βάλουμε μετά το α. Οπότε νομίζω ότι πάμε προς σωστή κατεύθυνση και αυτό είναι καλό για τον καταναλωτή και οπωσδήποτε υποστηρίζω την αλλαγή για να πάμε σε κατηγορίες α έως g. Από την άλλη πρέπει και ο έλεγχος της εφαρμογής ε, να γίνει πιο σοβαρός και βεβαίως τίθεται το ερώτημα του εάν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η σήμανση. Βουλεύτης ε, Μάριας, Μάριας. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική της ενεργειακής απόδοσης βρίσκεται σε συνάρτηση με αποφάσεις που αφορούν τους τομείς της ασφάλειας εφοδιασμού, της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, έτσι όπως έχει η κατάσταση σήμερα, ειδικά στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου είναι σημαντικό η ενεργειακή απόδοση να στοχεύει πρωτίστως στην εξάλληψη του ντροπιαστικού φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας. ο στόχος που έθεσε το συμβούλιο της ευρωπαϊκής ένωσης τον οκτώβριο του 2014 είναι η αύξηση στο 27% της ενεργειακής απόδοσης έως το 2030. Για να γίνει αυτό θα πρέπει οι πάροχοι και πολιτές σε όλα τα κράτη-μέλη να παρέχουν έγκυρες και ορατέ πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων τους πρέπει να αποφευχθεί η σύγχυση των καταναλωτών αλλά και να επιτευχθεί μια μετάβαση κατευθυνόμενη από τη γνώση. η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μπορεί να δώσει ένα ισχυρό κίνητρο τόσο στα κράτη μέλη όσο και στους ίδιους τους πολίτες να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή εξοικονόμησης ενέργειας και η επιτροπή θα πρέπει να βρει τους αναγκαίους πόρους για να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Ιβαν Ιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την στήριξή μου προς την έκθεση αυτή που πιστεύω ότι θα συμβάλλει και εξυπηρετώντας τους ε, παραγωγούς των διαφόρων προϊόντων αλλά θα εξυπηρετήσει και τους καταναλωτές. Μας μπερδεύει κάπως ε, αυτή η αναφορά της ε, ενεργειακής απόδοσης. Απλά, με απλά λόγια για να καταλαβαίνει ο κόσμος θα πρέπει να τα πούμε απλά και ξεκάθαρα και γι' αυτό είμαι υπέρ της έκθεσης. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν μπορούμε σε μια ενιαία αγορά να σκεφτούμε και άλλα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες ε, και να βρούμε ένα απλό και κατανοητό σήμα για την ποιότητα των υπηρεσιών, για την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και για την ενεργειακή απόδοση. Επιτέλους αυτό χρειαζόμαστε και θέλουμε ενοποιημένο τρόπο χαρακτηρισμού της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Last but not least, ο κύριος Κέλλη. Παρακολούθησα την COP21 στο Παρίσι και καταλήξαμε σε μια καλή σχετικά συμφωνία. Τώρα προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη μείωση των διοξιδίων των αερίων του θερμοκηπίου και να αναχαιτήσουμε την ε, αύξηση της ε, θέρμασης του πλανήτη, να μην ξεπεράσουμε τους 1,5 βαθμούς. Και η ενεργειακή απόδοση θα συμβάλλει σε αυτό το σκοπό. Έχουμε στόχους, τώρα αρχίζουμε και συζητούμε τις λεπτομέρειες. Ιδιαίτερα θέλουμε να προστατεριστούμε τους καταναλωτές, αυτούς που θέλουν να συμβάλλουν, που θέλουν να σώσουν τον πλανήτη και που φυσικά να μειώσουν τους λογαριασμούς που πληρώνουν για προϊόντα ενέργειας. Και δεν είναι τι θυσίμα θα βρούμε αν θα είναι ε, μεσίνη με άλλο τρόπο. Το θέμα είναι να έχουμε μια καλύτερη, απλούστερη ταξινόμηση της ενεργειακής απόδοσης ε, για να την καταλαβαίνει καλύτερα ο πολίτης και να συμβάλλει και αυτός στην υλοποίηση αυτών των αξιέπαινων στόχων. Ευχαριστώ. Εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα, η Επίτροπο Σεσίλια Μάλμστρομ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ευχαριστώ για τη χρήσιμη συζήτηση. Υπάρχει ισχυρή συνένεση και μεγάλη υποστήριξη για την αναθεώρηση του σήματος ε, απόδοσης για να είναι πιο χρήσιμο και βολικό για τον καταναλωτή. Για τη βάση δεδομένων δεν θα είναι μεγάλο φορτίο διοικητικό. Ε, δημιουργεί την ανάγκη μόνο καταχώρησης του μοντέλου ανεβάζοντας πληροφορίες που ήδη απαιτούνται με βάση τις ε, διάφορες κατεξουσιοδότης πράξη. Η τεχνική, η τεχνική τεκμηρίωση θα ε, δίνεται στις ε, αρχές εποπτείας της αγοράς, επιτήρησης, οπότε θα είναι σίγουρες πληροφορίες. Η Επιτροπή έχει εμπειρία με τέτοιες βάσεις δεδομένων από τα καλλιντικά και το κόστος θα μπορούσε να είναι και μικρότερο από το τωρινό. Γιατί οι κατασκευαστές δεν χρειάζεται να τηρούν τεχνική τεκμηρίωση για πέντε χρόνια για τις αρχές επιτήρησης της αγοράς μετά την τελευταία κατασκευή προϊόντος. Οπότε αυτό θα είναι χρήσιμο και δεν θα είναι πρόσθετο φορτίο για τους καταναλωτές. Συμφωνώ βέβαια ότι χρειαζόμαστε απλούστερα πρότυπα ε, καλύτερα για ολόκληρη την ε, εσωτερική αγορά. Δεν, θα μπορούμε να, δεν μπορούμε να το λύσουμε σήμερα το πρόβλημα, πάντως μπορούμε να στείλουμε ισχυρό μήνυμα ότι συμφωνούμε να κάνουμε κάτι σημαντικό για να διευκολύνουμε τους καταναλωτές να κάνουμε σημαντική δουλειά εδώ στην αναθεώρηση της σήμανσης ε, για την ε, ενεργειακή απόδοση και η Κομισιόν προσβλέπει στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να οριστικοποιήσει αυτή την πρόταση και ευχαριστούμε και τον εισηγητή και τους άλλους σκιώδεις για το έργο που έκαναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το είπα και στα Σουηδικά. Τώρα περνάμε στον εισηγητή μας, τον Τάριο Ταμπουράνο, παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο και όλους τους συναδέλφους για αυτή την διαδρομή που κάναμε μαζί, για τα μπράβο τους αλλά και για τις επικρίσεις που είναι και αυτές χρήσιμες ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα κείμενο ε, ισορροπημένο τελευταίου μήνες Ασχολούμαι με αυτή την έκθεση και όσο την ε, συνέτασα είχαμε και διαπραγματεύσεις και στο μυαλό μου είχα ένα όνειρο, είχα μια εικόνα το να υπάρχει αυτή η ετικέτα, η επισήμανση 2,0 2,0 όπως λέμε για να έχουμε μια αλλαγή οπότε δηλαδή αυτό φαντάστηκα ότι μια μέρα και εγώ ο ίδιος θα μπορούσα να μπω σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και να δω αυτή την ετικέτα. Αυτή που να ισχύει και να μπορούν όλοι οι Ευρωπαίοι να μπορούν να το κάνουν αυτό όπως το κάνανε κάποτε εδώ και χρόνια οι, οι Αυστραλοί και θα μπορούσαν να το κάνουν και διαβάζοντας, σκανάροντας με το κινητό οπότε έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτό όχι επί τη βάση μόνο των προκαθορισμένων χαρακτηριστικών να μπορούν επομένως ε, να έχουν κάτι σαν εφαρμογή που να μπορεί να τους βοηθήσει και να έχουν τις πληροφορίες. Ε, τις πληροφορίες που τους λένε ακριβώς ποιο είναι το πραγματικό κόστος η δαπάνη της συσκευής. Οπότε να μπορούν να επιλέξουν την συσκευή η οποία αντιστοιχεί περισσότερο στις ανάγκες τους και έτσι τελικά να ε, ε, έχουμε επενδύσει στις πιο αποτελεσματικές ε, συγκεκριμένες. Αυτό είχα στο μυαλό μου σε σχέση με την ετικέτα αυτή και ελπίζω το στιμότερο δυνατόν αυτό να συμβεί στον πραγματικό κόσμο μια που σήμερα η Ευρώπη χρειάζεται μια επιτυχία ένα success story. Έτσι ελπίζω να προχωρήσουμε από κοινού. Σας ευχαριστώ εγώ, λέει ο πρόεδρος, κύριε Ταμπουράνο. Σας ευχαριστούμε κύριε Ευρωβουλευτά. Ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψηφοφορία της έκθεσης Ταμπουράνο θα γίνει μεθαύριο ημέρα.